Σύμφωνα με την ε, ημερήσια διάταξη προχωρούμε στη σύσταση για δεύτερη ανάγνωση ως προς την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους ε, καταναλωτές. Και δίνω το λόγο στην εισηγήτρια για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, μετά από τρία χρόνια εντατικών εργασιών, μετά από πάνω από 3.000 τροπολογίες και άπειρες συζητήσεις, συνομιλίες, αντιπαραθέσεις, μετά από δύσκολες ε, τεχνικές ε, διαπραγματεύσεις και ε, τριμερή διάλογο, είναι τώρα για να ψηφιστεί το πολιτικό πακέτο μεταξύ των θεσμικών οργάνων για την επισήμανση των τροφίμων. Έτσι ο καταναλωτής θα παίρνει καλύτερες πληροφορίες για τα τρόφιμα, για στοχευμένη αγορά. Και όχι μόνο. Και οι κατασκευαστές τροφίμων θα βελτιωθούν με λιγότερη γραφειοκρατία, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Αυτό είναι σημαντικό ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πρέπει να ξέρουμε ότι ο τομέας των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται ε, στο πάνω από 80% από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η επισήμανση θα πρέπει να γίνεται για κάθε τρόφιμο από τα βασικά μέχρι τα πολύ επεξεργασμένα έτοιμα τρόφιμα. Γι' αυτό χρειάζεται, ε, δεν γίνεται υποχρεωτική επισήμανση με τα πρωτοκαλί κόκκινο-πράσινο. Ε, παρά τις δυσκολίες όμως, παρά τις ιδεολογικές πολιτικές αντιπαραθέσεις στο Κοινοβούλιο παρά τους εθνικούς εγωισμούς των κρατών μελών τώρα υπάρχει μια συμβαστική λύση τα αλλεργιογόνα έχουν πρώτη θέση φυτική προέλευση φυτικών ελαίων αναφέρεται Επίσης υπάρχει σήμανση καταγωγής για τα πουλερικά, για τα εγωπρόβια κρέατα, το χοιρινό. Ε, για άλλα θα, δείξω, θα δείξει αν θα προσθεθεί η καταγωγή για το γάλα και τα γαλακτοκομικά, ε, single ingredient ε, προϊόντα από ένα συστατικό, κρέας επεξεργασμένα, μεταποιημένα τρόφιμα κλπ. Ε, οι απομιμήσεις ε, θα αναφέρονται επίσης ξεκάθαρα μπροστά. Το ίδιο ισχύει για ε, κρέας που αποτελείται από μικρά κομμάτια. δεν θα πρέπει η επισήμανση, η συσκευασία να δίνει την εντύπωση ότι εκεί μέσα υπάρχει κάτι που δεν είναι. αν αναφέρονται φρούτα μέσα στο γιαούρτι πρέπει να υπάρχουν φρούτα όντως, όχι μόνο αρωματικά και ε, χρώματα. Είναι σημαντικό να δείχνουμε ανά 100 γραμμάρια ή μιλιλίτρα, να δείχνουμε την περιεκτικότητα για να υπάρχει συγκρισιμότητα. Ε, στο ψάρι και στο κρέας η ημερομηνία της πρώτης κατάψυξης και άλλα σημαντικά και όλα πρέπει να είναι ευανάγνωστα. Ε, έχω μπορεί στην αναγνωσιμότητα, την ευανάγνωστο και αναθέσαμε στην Κομισιόν να ορίσει δεσμευτικούς κανόνες για την αντίθεση δηλαδή μεταξύ της γραφής και της, του φόντου. Επίσης ε, πιστεύουμε ότι πρέπει να μειωθεί το κόστος και η γραφειοκρατία. Ε, πρέπει να υπάρχουν στοιχεία για τα αλλεργιογόνα ε, όταν είναι κατασκευασμένα τα τρόφιμα, προπαρασκευασμένα. Ε, υπάρχουν διάφορες ιδιαιτερότητες ε, που πρέπει να ληφθούν υπόψη και τις ε, διατηρήσαμε. Τώρα συμφωνήσαμε όλοι και οι ναι, σοβαροί συνομιλητές ικανοποιημένοι. Ευχαριστώ και τους σκιώδεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαίτερα τον Επίτροπο Τάλη για τις δηλώσεις που ελπίζουμε ότι θα κάνει και έτσι θα λύσει το γόρδιο δεσμό που είχαμε να αντιμετωπίσουμε στην πολιτική συζήτηση. Επίσης ευχαριστώ την Ουγγρική Προεδρία του Συμβουλίου που κατάφερε κάτι απροσδόκητο πραγματικά. Μπόρεσε σχεδόν να τετραγωνίσει τον κύκλο ε, χάνοντας μια συμφωνία στο ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο Υπουργός Σαβίνσκι έχει το λόγο από το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, με μεγάλη ευχαρίστηση παίρνω μέρος σήμερα στη σημερινή συζήτηση που καταλήγει μετά από τέσσερα χρόνια συζητήσεων για το θέμα της πληροφόρησης τον τροφή που δίνουν τα τρόφιμα στους καταναλωτές. Οι συζητήσεις υπήρξαν δύσκολες, αλλά το αποτέλεσμα αξίζει, άξιζε τις προσπάθειες αυτές. Ο κανονισμός φέρνει στους καταναλωτές και καταναλώτριες πολλά ωφέλη. Είναι σημαντικό βήμα για την εγγύηση του ότι τα τρόφιμα που αγοράζονται και καταναλώνονται στην Ένωση θα πολλούνται με βάση αξιόπιστες πληροφορίες στη συσκευασία. Οι διαπραγματεύσεις μας επέτυχαν λόγω της επικοδομητικής τάσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την εισηγήτρια, την κυρία Ρενάτα Ζόμερ και τους συνεισηγητές της, καθώς και όλους όσους συνεισέφεραν στην σημερινή κατάληξη της διαδικασίας. Ευχαριστώ και την προηγούμενε τις προηγούμενες προεδρίες. Έξι χρειάστηκαν να ασχοληθούν με αυτό το θέμα για να καταλήξουμε στη συμβιβαστική πρόταση που έχουμε σήμερα μπροστά μας και που ελπίζω να εγκριθεί αύριο. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι ο κανονισμός θα, αυτός θα διασφαλίσει στους καταναλωτές και καταναλώτριες πιο αξιόπιστες πληροφορίες που να λάβουν υπόψη την διατροφή τους χωρίς ταυτόχρονα να επιβαρύνει τις επιχειρήσεις. Και τα τρία όργανα κατέληξαν στο συμβιβασμό αυτό στα κυριότερα θέματα. Οι ετικέτες θα είναι σαφέστερες και καθαρότερες τα συσκευασμένα προϊόντα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν πληροφορίες για τις θερμίδες που περιέχουν και υποχρεωτικά θα αναφέρεται αν υπάρχουν αλλεργιογόνα. Τα τρόφιμα που θα πολλούνται χωρίς συσκευασία θα τους εφαρμόζεται ειδική. Θα τους εφαρμόζονται ειδικέ διατάξεις και για να μην επιβαρυνθούν πολύ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις ετικέτες, της συσκευασίες, τα μη συσκευασμένα προϊόντα ή εκείνα που παράγουν μικρές εταιρείες εξαιρούνται από την υποχρεωτική αυτή πληροφόρηση. Όλη η πληροφόρηση θα πρέπει να χορηγείται πριν, να είναι διαθέσιμη πριν τη στιγμή της αγοράς. Επίσης υπήρξαν συμβιβασμοί σε τρία άλλα θέματα για τη συσκευασία τα οποία ακόμη επεξεργάζεται η Κομισιόν. Είναι τα είναι η χώρα προέλευσης και η δήλωση των πληροφοριών για την παρουσία Transfats. Η Κομισιόν μας υπέβαλε έκθεση, τα υποβάλλει έκθεση για την πρόοδο και την επιτυχία της πολιτικής αυτής μετά από τρία χρόνια. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να έχει και άλλα δικά της νομοθετικά συμπεράσματα. Κυρίες και κύριοι, ο κανονισμός αυτός αποφέρει πολλά ωφέλη στους καταναλωτές και καταναλώτριες, αυξάνει τη διαφάνεια και εφόσον θα είναι πιο απλές οι ετικέτες τώρα, θα μας βοηθάει επίσης να εφαρμόσουμε σωστότερα τον Ευρωπαϊκό Νόμο. Θα αρχίσει, ελπίζουμε, να εφαρμόζεται όσο το δυνατόν συντομότερα, αφού εξακριβώσουν οι δικηγόροι την ε, κατά πόσον είναι εφαρμόσιμο θα αρχίσει να εφαρμόζεται και θα δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα ελπίζουμε πριν τα τέλη του Οκτωβρίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Υπουργό. Ο Επίτροπος Νταλή έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη Τρία χρόνια πριν, στις 30 Ιανουαρίου 2008, η Επιτροπή ενέκρινε μία πρόταση κανονισμού για πλήρη πληροφόρηση των καταναλωτών. Τώρα φτάνει στο πέρας αυτή η διαδικασία έγκρισης του κανονισμού. Θα ήθελα να πω ότι είμαι ευγνώμη προς την κυρία Ζόμερ γιατί επιτέλεσε πολύ σκληρή εργασία για να φτάσουμε σε συμβασμό με το Συμβούλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους σκιώδεις. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ουγγρική Προεδρία και τις προηγούμενες προεδρίες που ήταν ιδιαίτερα δραστήριες έτσι ώστε να εξεύρουμε συμβιβασμούς που να γίνουν αποδεκτοί από το Συμβούλιο. Χαίρομαι διότι το Κοινοβούλιο συμμερίζεται το, την θέση μας έτσι ώστε να έχουμε μια γενικότερη πλαισίωση πληροφόρησης για τους καταναλωτές, όπου οι καταναλωτές να έχουν την πρώτη θέση. Πρόκειται για, έναν, ε, για ένα ευέλικτο πλαίσιο που θα ανταποκριθεί και σε μελλοντικές εξελίξεις. Η κοινή μας εργασία κατά τους προηγούμενους μήνες ε, ανταμείφθηκε σε πολλούς τομείς. Καταρχήν, υπάρχει ένα ελάχιστο όρο, ε, ε, όριο υποχρεωτικής πληροφόρησης. Εδώ υπήρχαν πολλά παράπονα υποχρεωτικές πληροφορίες για τη διατροφική αξία έτσι ώστε να αναγνωρίζουν οι καταναλωτές τα, τα προϊόντα ανάλογα με τις διατροφικές τους συνήθειες. Επίσης, αλλεργιογόνες ουσίες όχι μόνο στα προσυσκευασμένα αλλά και στα μη προσυσκευασμένα προϊόντα έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη προστασία. Επίσης θα πρέπει να ορίζονται τα αλλεργιαγόνα επακριβώς για να τα αναγνωρίζει ο καταναλωτής. Η υποχρεωτική σήμανση αυτή θα ε, εξασφαλίσει το ότι οι καταναλωτές θα έχουν σκόπιμες και χρήσιμες πληροφορίες. Ο Επίτροπος Τσόλος, ο συνάδελφός μου που είναι υπεύθυνο για τη Γεωργία και εγώ προσδίδουμε μεγάλη σημασία σε αυτό το τομέα. Αυτό βοηθά και τους ε, καταναλωτές, αλλά ε, λυπάμαι διότι βλέπω ότι ένα μεγάλο μέρος της αρχικής πρότασης Επιτροπής έχει διαγραφεί. Αυτό μειώνει το ευεργέτημα της συμπερίληψης ε, διατροφικών πληροφοριών στο μπροστινό μέρος της συσκεσίας. Αυτό αποτελεί όμως ένα βασικό ε, βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Επίσης, λυπάμαι διότι τα αλκοολούχα ε, δεν υποβάλλονται σε αυτή την υποχρέωση σήμανσης ως προς τα συστατικά. Ο καταναλωτής πρέπει να λαμβάνει αυτές τις πληροφορίες όταν καταναλώνει αλκοολούχα ποτά και θα πρέπει να μπορούμε να βρούμε όλα αυτά τα στοιχεία στη σήμανση. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και πληροφόρηση επιτροπής ως προς την σφαγή των ζώων γιατί οι καταναλωτές προσδίδουν μεγάλη σημασία σε αυτό, δηλαδή κατά πόσο τηρούνται οι κανόνες τη στιγμή της φαγής. Επίσης γνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγάλη ευαισθησία ως προς αυτό το θέμα. Έχει γίνει μία μελέτη έτσι ώστε να δίδονται αυτές οι πληροφορίες σε σχέση με τον ε, τρόπο σφαγής. Δεύτερον, υπάρχει μία δήλωση της Επιτροπής για την Ασπαρτάμι. Η ΕΦΣΑ θα προβεί σε μία νέα αποτίμηση της ασφάλειας της ασπαρτάμις. Η ΕΦΣΑ δέχτηκε αυτό το αίτημα και θεωρούμε ότι η αξιολόγηση θα λήξει το Σεπτέμβριο του 2012. Η Ευρωπαϊκή Αρχή επίσης θα ασχοληθεί, για την ασφάλεια των τροφίμων θα ασχοληθεί και με την ασπαρτάμι όταν την λαμβάνουν οι έγκυες γυναίκες. Επίσης θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ως προς τα ανώτατα επιτρεπτά ποσά και πληροφορίες προς τους καταναλωτές. Τρίτον, ως προς τις θερμίδες στα τρόφιμα, ζητάμε πληροφορίες σε ε, σχέση με για εκχυλίσματα τροφίμων και τη θερμιδική τους αξία. Έτσι θα μπορέσουμε να δούμε τι γίνεται και στην περίπτωση χρήσης χρωστικών ουσιών στα τρόφιμα. Τέταρτον, μία δήλωση της Επιτροπής ως προς τον προσυσκευασμένων για άμεση πώληση προϊόντων και τις προαπαιτήσεις υγείας, τα προαπαιτούμενα υγείας. Αυτό έχει σχέση και με το πακέτο υγείας και υγιεινής. Τέλος, θα ήθελα να κάνω το εξής, την εξής δήλωση. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι αντιτίθεται στον κανονισμό 182 κάθετος 11 είναι αντίθετο το να, το να ε, ψηφιστεί το άρθρο 5.2.1β. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει η Επιτροπή να ορίσει μία εφαρμοστική πράξη εκεί που θεωρείται αναγκαίο. Επειδή πρόκειται για τη χρήση του 5-4 και ε, ως προς το 5-2 δεν πρόκειται για διεκριτική ευχέρεια του νομοθέτη, αλλά θα πρέπει να ερμηνευθεί συσταλτικά αυτή η διάταξη. Ναι, ναι. Το πακέτο συμβιβασμού αποτελεί ένα βασικό βήμα στον τομέα της πληροφόρησης ως προς τις τροφές και τη διατροφική, τα διατροφικά συστατικά. Τώρα το λόγο έχουν οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Λίζε για δύο λεπτά από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θερμά συγχαρητήρια καταρχήν στην εισηγήτρια Ρενάτε Ζόμερ, ευχαριστίες σε όλους όσους βοήθησαν, συμπεριλαμβανομένου του Επιτρόπου Τζον Ντάλι και της Ουγγρικής Προεδρίας. Την νομοθετική διαδικασία την παρακολούθησα από την αρχή, πράγματι ήταν δύσκολη με διαφορετικές θέσεις, διαφορετικά συμφέροντα, αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι καλό. Ε, ο καταναλωτής ε, έτσι θα έχει από μας καλύτερες, σαφέστερες πληροφορίες δεν θα κυδεμονεύουμε όμως τον καταναλωτή και δεν θα του υπαγορεύουμε τι θα τρώει και τι δεν θα τρώει. Τονίζω ιδιαίτερα τη συμφωνία για τις απομιμήσεις. Για μας ε, ήταν πολύ σημαντικό πάντα στην ομάδα μας ε, τα τρόφιμα να μην δημιουργούν την εντύπωση ότι αποτελούνται από ένα βασικό τρόφιμο ενώ αυτό δεν είναι αλήθεια. Με άλλα λόγια, ε, προϊόντα γάλακτος ας πούμε ε, θα πρέπει να αναφέρεται αν υπάρχει δεν υπάρχει γάλα ή αν υπάρχουν, τι έλαια ε, περιλαμβάνει ένα προϊόν. Ε, αν αναφέρεται απομίμηση μπορεί η εταιρεία να πει όχι δεν είναι απομίμηση είναι καινοτόμο προϊόν. Όταν όμως γράψουμε και τα συστατικά τα οποία συνήθως δεν περιλαμβάνονται ενώ τώρα θα, θα περιλαμβάνονται ε, αυτό αποτελεί μεγάλη βελτίωση. Οι καταναλωτές δεν θα παραπλανώνται πια από, τα, από τις απομιμήσεις τροφίμων και η παραγωγή θα, για παράδειγμα γάλακτος θα επιτυγχάνουν καλύτερες τιμές στα προϊόντα τους. Ε, βέβαια δεν χρειάζεται μεγεθυντικός φακός, ε, δεν πρέπει να χρειάζεται μεγεθυντικός φακός για να διαβάσουμε τι λέει και επίσης ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τι μπορούν να κάνουν. Μην έχουμε υπόψη μας μόνο την Εστλέ Φεραίρο και άλλοι και ο μικρός αρτοποιός και ο μικρός εστιάτορας θα πρέπει να μπορούν να τα βγάζουν πέρα ή αυτός που πουλάει ε, τα προϊόντα του από την εκμετάλλευση. Ευχαριστούμε θερμά και θερμά συγχαρητήρια. Εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η κυρία Βίλμοτ για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι γιατί μετά από τόσα χρόνια εργασία κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση πληροφορώντα του καταναλωτέ και καταναλώτριε τι περιέχουν τα τρόφιμα που καταναλώνουν. Δυστυχώ φαίνεται σαν να ξεχάσαμε ότι πρόκειται για πληροφόρηση των καταναλωτών ακριβώς οι πιέσεις που άσκησαν τα διάφορα λόμπι ήταν εντυπωσιακέ. Προσπάθησαν να σταματήσουν τη διαφανή ετικετοποίηση. Πάντως υπάρχει αυτός ο συμβιβασμός και χαίρομαι που το Συμβούλιο δέχτηκε να αναφέρεται η χώρα προέλευσης για ορισμένα τουλάχιστον προϊόντα κρεάτων. Επίσης πείσαμε το Συμβούλιο ότι πρέπει Κομισιόν να κάνει μία έκθεση για την προέλευση των μεταποιημένων κρεάτων. Αυτή τη στιγμή μπορώ να αγοράσω ένα συσκευασμένο σάντουιτς με κοτόπουλο που να λέει ότι παρήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο ενώ το κοτόπουλο είναι από το Ταϊβάν. Τα πρόσθετα στοιχεία που δίνονται στα τρόφιμα μπορούν καμιά φορά να δημιουργήσουν ιδίω τα υδρογονωμένα λίπη και καρδιακές παθήσεις. Γι' αυτό πρέπει να κάνει νέα εξέταση σε τρία χρόνια η Κομισιόν και να απαγορευθούν τα πρόσθετα αυτά υδρογονωμένα λίπη όπως γίνεται στην Αυστρία και τη Δανία. Επίσης όλα τα λάδια πρέπει να αναφέρεται η σύστασή τους για να πιεστούν οι κατασκευαστές να χρησιμοποιούν έλαια από βιώσιμες πηγές. Δυστυχώς βέβαια δεν, έχει γίνει δεν έχουν γίνει δεκτές όλες οι προτάσεις μας, που μερικές από τις οποίες θα συνέβαλαν στην καταπολέμηση σοβαρών ασθενειών όπως την καρδιοαγγειακές και το διαβήτη. Παρ' όλα αυτά χαίρομαι γιατί μπορούν εθελοντικά να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται συστήματα που έχουν αποδείξει την επιτυχία τους. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι πρώτη φορά που θα είναι υποχρεωτική η πληροφόρηση για τα τρόφιμα από τον ενωσιακό νόμο. Θα βλέπει κανείς πόσο αλάτι περιέχεται παραδείγματος χάρη σε ένα συσκευασμένο τρόφιμο. Είναι λοιπόν μια πρόοδος, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για περισσότερες πρόοδους υπέρ των καταναλωτών και καταναλωτριών. Ευχαριστούμε. Από τους ε, φιλελευθέρους, για ένα λεπτό, ο κύριος Γκέρμπραντ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Ζόμερ, του Σκιώδη, την Ουγγρική Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα επίσης ε, να τους ε, ευχαριστήσω γιατί καταφέραμε πολλά για 700 εκατομμύρια καταναλωτές για να γνωρίζουν τι περιέχει η διατροφή τους. Επίσης, δεν επιβάλλουμε στους καταναλωτές τι θα καταναλώνουν, Απλώς θα τους δίνουμε πληροφορίες έτσι ώστε να μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα. Αυτό δεν αρκεί. Θα πρέπει και στα σχόλια να προσδώσουμε μεγαλύτερη σημασία στην υγιή διατροφή. Επίσης, θα πρέπει να μιλάμε για φυτικά έλαια στην σήμανση. Θα πρέπει να υπάρχει αυτή η σήμανση έτσι ώστε να ε, μην μπορεί να γίνει χρήση των ακορέστων. Νομίζω ότι με αυτό το συμβιβασμό θα φτάσουμε σε μία μεγάλη πρόοδο ως προς τα λύπη. Είδα ότι ότι ο Επίτροπος διαβάζει το iPad του. Δεν ξέρω κατά πόσο στο μέλλον δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε νέες τεχνολογίες για να ε, μπορούμε να δίνουμε πληροφορίες και προς τους καταναλωτές για να μην βασίζονται στην σήμανση επιχάρτου. Ο κύριος Σλούτερ για δύο λεπτά από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις καταφέραμε κάτι καλύτερο. Παρόλο που χάθηκε μια ευκαιρία για γρήγορη διαδικασία. Επίσης το λόμπι για του, του έβγαλε τα αλκοολούχα. Πόσοι ξέρουμε για τις επιπτώσεις της μέθης. Πολύ. Πόσοι όμως ξέρουμε πόσες θερμίδες έχει ένα ποτό. Έχουμε δικαίωμα να τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ χαίρομαι διότι μειώνονται οι δυνατότητες ε, απάτης από το σύστημα αυτό θα ξέρουμε με το ζαμπόν στο σάντουιτς ε, από τι αποτελείται, αν αποτελείται από κρέας ολόκληρο κομμάτι ή από κομμάτια σχηματισμένο, δηλαδή από πολλά κομμάτια κρέας ε, και το ίδιο ισχύει και για πολλά άλλα τρόφιμα. Ε, επίσης τα φυτικά έλεα θα αναφέρονται, καλό αυτό. Και η επισήμανση του κρέατος θα αρχίσει να γίνεται πολύ πιο, με πολύ πιο διευρυμένο τρόπο και καταναλωτές που θέλουν να αποφεύγουν κάποια είδη κρεάτων και θέλουν να ε, προτιμήσουν ε, αυτούς που τα παράγουν κατά από καλές ε, συνθήκες θα μπορούν να το κάνουν. Τα τρανσλιπαρά θα αναφέρονται επίσης. Δεν είχατε συμφωνήσει με την απόφαση του Κοινοβουλίου, αλλά τουλάχιστον θα διεξαχθεί μελέτη. Και μπορεί έτσι να ε, παίξουμε ένα ρόλο με την επισήμανση να μειωθούν οι καρδιοπάθειες και να βοηθήσουμε και με την επισήμανση των αλλεργιογόνων. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν όλο αυτό. Από τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές, ο κύριος Στίβενσον, για ένα λεπτό. Πρόεδρε, χαίρομαι γιατί το Συμβούλιο, Επιτροπή και Κοινοβούλιο φτάσαν σε μία συνένεση. Υπήρχε μεγάλη διχογνωμία, αλλά εργαστήκαμε για τρία χρόνια και θα θέλαμε να συγχαρούμε τη Ρενάτ Σόμερ. Θα ήταν κρίμα να μην επιτύχουμε όπως έγινε με τα νέα τρόφιμα. Όπως είπε και ο κύριος ε, Νταλή, μίλησε για τα σφαγιαστέντα ζώα, στα οποία δεν γίνεται μία ένεση ανεσυτοποίησης όταν μιλάμε ιδιαίτερα για κρέας χαλάλ. Αυτό οδήγησε σε μεγάλες κατάχρησεις, δηλαδή η εξαίρεση έτυχε κατάχρησης και έτσι σφαγιάζονται τα ζώα κατά αυτόν τον τρόπο και μετά μπαίνουν στη διατροφική αλυσίδα. Οι καταναλωτές στην Ευρώπη πρέπει να γνωρίζουν όταν αγοράζουν αυτά τα προϊόντα. Ο κύριος Ντάλι είπε ότι θα προωθήσει έναν κανονισμό για την ευζοία των ζώων και αυτό ακριβώς περιμένουμε από εκείνον. Από πλευράς ε, Γκουε, η κυρία Λιωτάρ, για 1,5 λεπτό. Κύριε Ντάλη, έχω ένα δώρο για σας. Σήμερα γιορτάζουμε το πρόβατο Ντόλι, όχι Ντάλι αλλά Ντόλι, το πρώτο κλωνοποιημένο ζώο το οποίο όμως πέθανε το 2003 Παρόλα αυτά, αυτό δείχνει ότι όλα τα κλωνοποιημένα ζώα μέχρι τώρα ζουν πολύ λίγο. Δεν ξέρω αν πρέπει να χαρούμε λοιπόν για αυτή την, ε, αυτό το κατόρθωμα. Τουλάχιστον η Κομισιόν μπορούμε να πούμε ότι 15 χρόνια χρειάστηκε για να εγκρίνει κάποια νομοθεσία για τα γενετικώς τροποποιημένα, για να μην εγκρίνει νομοθεσία για τα γενετικώς τροποποιημένα ζώα και θα συνεχίσει η εμπορία τους χωρίς να το γνωρίζει ο καταναλωτής ούτε η καταναλώτρια. Τι θα λέει η ετικέτα για αυτά τα ζώα, τίποτα. Και τα πολυακόρεστα που βλάπτουν την υγεία επίσης δεν θα αναφέρονται τίποτα. Η προέλευση τώρα, μόνο για το φρέσκο κρέας, όχι για το συσκευασμένο. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά που κάναμε και πριν χωρίς χρήσιμες πληροφορίες για τον καταναλωτή και την καταναλώτρια για τη ζάχαρη, το αλάτι κτλ. Τέλος η Ευρώπη επέλεξε τα κρέατα που τα ζώα που σφάζονται χωρίς τον ενομισμένο τρόπο να μην αναφέρεται αυτό. Εδώ πάλι ξεγελιέται ο καταναλωτής και η καταναλώτρια. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή την ημέρα που σε εισαγωγικά γιορτάζουμε την ε, δημιουργία της Ντόλη δεν έχουμε λόγο να χαιρόμαστε. Το λόγο είχε ο κύριος ε, Ρώση από την Ευρώπη της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας. Ήμασταν υπέρ του κειμένου στην πρώτη ανάγνωση. Το Συμβούλιο όμως απέρριψε το κείμενο που βρίσκεται τώρα σε δεύτερη ανάγνωση, διότι στη σήμανση δήθεν δεν πρέπει να φέρεται η χώρα προέλευσης. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η επιλογή αντιτάσσεται στα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας. Στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Επιτροπής και Συμβουλίου έγινε ένα βήμα προς τα μπρος, αλλά είναι πολύ περιορισμένο σε σχέση με τις απαιτήσει των Ευρωπαίων πολιτών. Θα πρέπει να υπάρχουν εθνικές διατάξεις που να μην παραμένουν κενό γράμμα. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι μέσα στο πλαίσιο της ε, μόνιμης επιτροπής χρειάζεται η ειδική πλειοψηφία. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζει ο καταναλωτής με τι διατρέφεται και ακριβώς αυτό υποστηρίζουμε και εμείς. Εξ των μη εγγεγραμμένων, ντότς για ένα λεπτό. Thank you. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, ευχαριστώ την εισηγήτρια. Οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα για σωστή και όχι παραπλανητική επισήμανση. Η διατροφική ενημέρωση είναι σημαντική και τα ποιοτικά πρότυπα των τροφίμων είναι σημαντικά για την επιλογή και την ασφάλεια των καταναλωτών. Όλα αυτά είναι καλά πράγματα και πραγματικά προέκυψαν από την έκθεση. Θέλω όμως να υπογραμμίσω έναν τομέα ειδικότερα που με απασχολεί και αφορά ε, την χώρα προέλευσης και την ένδειξη τη σχετική. Έχω επιφυλάξει σε σχέση με τον πιθανό αντίκτυπο στο εμπόριο στη Βόρεια Ιρλανδία οι τοπικές επιχειρήσεις ήδη ε, είδαν ότι οι ενδείξεις προέλευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προστατευτικό μέτρο με αρνητικό αντίκτυπο στο εμπόριο της Βορείου Ιρλανδίας και οι παραγωγοί και οι μεταποιητές ε, ζημίωσαν ως αποτέλεσμα. Ξέρω ότι αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το εξετάσουν και απασχολεί τα κράτη-μέλη. Εγώ θα καλούσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεξαγάγει μία μελέτη επιπτώσεων και να διερευνήσει τυχόν ε, προτινόμενη νομοθεσία επισήμανσης σχετικά με την αναφορά της ένδειξης προέλευσης. Ευχαριστώ. Το λόγο έχουν τώρα οι λοιποί εγγεγραμμένοι αγορητέ. Πρώτη η κυρία Γιούζο για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η κυρία Σόμερ και οι σκιώδεις ηγητές, η Ουγγρική Προεδρία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξαν σε μια καλή συμφωνία για τον κανονισμό αυτό. Σημαντικό και για τους καταναλωτέ και για την επιστημιστική ασφάλεια. Και πολλά συγχαρητήρια. Ως καταναλωτές είναι λογικό να θέλουμε εξαντλητική ενημέρωση και πληροφόρηση για ό,τι τρώμε. Αλλά δεν είναι καθόλου εύκολη αυτή η πληροφόρηση στις συσκευασίε. Γι' αυτό θα πρέπει να ζητήσουμε μια ισορροπία και μάλιστα ισορροπία με σχέση κόστους-οφέλους. Γιατί η πληροφορία στην ετικέτα κοστίζει και κάποιος θα πρέπει να πληρώνει αυτό το κόστος. Και αν δεν το πληρώνει ο καταναλωτή, σημαίνει ότι πολλέ μικρομεσαίε επιχειρήσει θα πρέπει να βγουν από την αγορά, γιατί δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τι μεγάλε, οι οποίε μπορούν να υπομισθούν το επιπλέον κόστο τη ετικέτα. Θα πρέπει λοιπόν πάντα να ζητούμε μια ισορροπία γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι Ε, πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι τελικά. Για την ετικέτα για τη χώρα προέλευσης είχε προβλεφθεί σε περίπτωση σύγχυσης να γράφεται στην ετικέτα η προέλευση των προϊόντων. Και σε ό,τι αφορά τα μεταποιημένα προϊόντα που έχουν πολλά συστατικά δεν είναι εύκολο να ε, καθορίσει κανείς ποιο είναι το βασικό συστατικό. Άρα Όλα αυτά έχουν προβλήματα, έχουν κόστος και διοικητική ε, επιβάρυνση και για τις ε, επιχειρήσεις χωρίς να είναι σαφές το πλεονέκτημα για τον καταναλωτή. Επιπλέον, σε αυτά τα πλαίσια συμφωνώ να μην ε, υπαχθούν εδώ τα εινοπνευματόδη γιατί ρυθμίζεται με τρόπο πάρα πολύ αυστηρό η ετικέτα τους. Και όλοι ξέρουν ότι το πνεύμα έχει και θερμίδες, δεν χρειάζεται να το γράφουμε τώρα επιπλέον. Είναι πολύ σημαντικό, αλλά πιο σημαντικό είναι η καλή ενημέρωση του καταναλωτού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, ευχαριστώ πολύ. Ε, Για 1,5 λεπτό δεκάστρο. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για ένα νέο και σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση του στόχου που είναι η προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστώ την εισηγήτρια, την κυρία Σόμερ και ευχαριστώ όλους τους σκιώδεις εισηγητές, ε, κυρία κυρίως την κυρία Κλένη Κουίκομ που είναι η σκιώδη εισηγήτρια της ομάδας μου ε, για να ε, έχουμε το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον με εμπιστοσύνη είναι αλήθεια ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η δεύτερη ανάγνωση αναθεωρεί αυτά τα οποία ελέγχθησαν στην πρώτη ανάγνωση. Παραδείγματο χάρη, θέλω να πω ότι εμεί περιμέναμε πολλά περισσότερα όσον αφορά την επισήμανση προέλευση των γεωργικών προϊόντων. Η υποχρέωση να αναφέρεται η προέλευση όλων των ε, ειδών κρέατο. Είναι μια πολύ σημαντική καινοτομία που ανταποκρίνεται στις προσδοκίε ε, των Ευρωπαίων καταναλωτών. Βεβαίως πρέπει να υπογραμμίσουμε και τις ε, πιο ε, χαμηλέ φιλοδοξίε όσον αφορά την υποχρεωτική επισήμανση για όλα τα νοπά αγροτικά προϊόντα και για τα μεταποιημένα συστατικά. Η ίδια η επισήμανση των, των ειδών αποκλείει ορισμένες σημαντικές παραγωγές που καθιστούν απαραίτητο υπάρχει άλλη μορφή προστασία όπως ε, το κρέας ε, κουνελιού, ε, Γι' αυτό λοιπόν ο δρόμος που πρέπει να ακολουθεί έχει ήδη χαραχθεί και τώρα πλέον είναι απαραίτητο να ακολουθήσουμε τον δρόμο αυτό με την ίδια δέσμευση και υπευθυνότητα που μας έφερε μέχρι εδώ. Ευχαριστούμε κύριε Τεκάστρο. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Ρίς. Ευχαριστώ. Μετά από τρία χρόνια συζητήσεων αρκετά σφοδρών τελικά αυτός ο κανονισμός ε, για τις πληροφορίες στους καταναλωτές ε, είναι έτοιμος ε, προς χρήση. Το θέμα της διευρυμένης μνήμης της χώρας προέλευσης ανταποκρίνεται σε σημαντική απέτηση των πολίτων να γνωρίζουν την προέλευση του προϊόντος ώστε να δώσουν έμφαση σε ντόπια προϊόντα, να αναφαίνονται ξεκάθαρα τα αλαριογόνα. Επίσης το θέμα της ασπαρτάμης που ζητήθηκε από την ΕΦΣΑ. Σε ό,τι αφορά τα τρανς λιπαρά, τα υδρογονοποιημένα βιομηχανικά ελίθη που, περιλαμβάνονται στα γλυκά, σε διάφορα προϊόντα που έχουν τηγανιστεί στις πίτσες. Ε, γνωρίζουμε ποια είναι τα ολέθρια αποτελέσματα αυτών των τρας λιπαρών. Γιατί δεν έδρασε πιο γρήγορα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν το καταλαβαίνω αυτό από όλοι. Δεν αρκεί μία απλή αναφορά των τρανς λιπαρών στην ετικέτα. Θα έπρεπε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση γιατί 300.000 ε, νέα κρούσματα παχυσαρκίας έχουμε στην Ευρώπη και θέλουμε να ε, καταπολεμήσουμε την παχυσαρκία με κάθε τρόπο. Δεν ξέρω γιατί δεν δόθηκε αρκετή έμφαση στα τρανς λιπαρά. Κυρία Γκέρλινγκ, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την δόκτωρα Ζόμερ και τους σκιώδης ηγητές γιατί φαίνεται ότι ανάγεται στο παρελθόν αυτό το θέμα. Εγώ μόνο στην τελευταία κοινοβουλευτική θητή ήμουν ευρωβουλευτή, αλλά για σας φαντάζομαι ε, θα τράβηξε πολύ αυτό το θέμα. Χαίρομαι για την περισσότερη διαφάνεια στην επισήμαση των ε, τροφίμων, γιατί έτσι αναγνωρίζονται τα συμφέροντα των καταναλωτών. Είχαμε εκατοντάδες χιλιάδες ε, παρατηρήσεις και παράπονα που μας έκαναν οι καταναλωτές και χαίρομαι γιατί και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις όπως αντίστοιχε στο Ηνωμένο Βασίλειο συμμετείχαν στην ενημερωτική εκστρατεία. Βέβαια δεν είναι απόλυτα ικανοποιητικό ο κανονισμό. Έχουμε ακόμη δρόμο να, δια... διανύσουμε, για παράδειγμα για τη μνήμα τη χώρα προέλευση, αλλά εδώ τουλάχιστον είναι αρκετά καλή συμβαστική λύση. Ό,τι αφορά τα στοιχεία τη θρεπτική αξία, θα πρέπει να είναι και εύχριστα και βανάγνωστα και τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν με την διακριτική τους ευχέρεια, αλλά να, να διασφαλιστεί η αναγνωσιμότητα των ετικετών. Νομίζω θα συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών αυτή η οδηγία και από αυτή την άποψη είναι πολύ καλή. Για ένα λεπτό το λόγο έχει ο κύριο Σκότα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο καταναλωτής είναι η λέξη κλειδί αυτής της έκθεσης και πολύ συχνά ξεχνάμε σε ποιον απευθυνόμεθα όταν λαμβάνουμε αποφάσεις. Για να υπάρχει λοιπόν καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή έχουν ληφθεί ή συζητούνται σημαντικά θέματα όπως παραδείγματος κάνει η συζητουνται σημαντικα θεματα οπως παραδειγματο κανει η ενδειξη της διατροφικής αξίας ή ε, της προέλευσης. Είναι σημαντικό το βήμα αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Η προέλευση για τα γεωργικά προϊόντα η ένδειξη των ε, σημαντικών συστατικών. Αυτή είναι η πρώτη πληροφορία που πρέπει να δίνουμε στον καταναλωτή. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις όπου η χνηλασιμότητα είναι καθοριστική σημασία. Ε, ε, πρόσφατα είδαμε ότι είχαμε ένα βακτήριο το οποίο στήξε τη ζωή πολλών ανθρώπων. εάν το γνωρίζαμε αυτό και αν το γνωρίζει κανείς μπορεί να αντιδράσει πολύ ταχύτερα. στον τομέα του, του ανταγωνισμού η, ονομασία, η προέλευση, η ένδειξη προέλευσης είναι συνώνυμο της ποιότητα. Και ορισμένε χώρε μπόρεσαν με τον τρόπο αυτό να αποκτήσουν, να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του καταναλωτή. Εμεί στηρίζουμε την ένδειξη τη προέλευση για να γνωρίζει και ο καταναλωτή τι ακριβώ καταναλώνει. Ευχαριστώ. Για ένα μισή λεπτό, κυρία Ντελαμή. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας φυσικά, ε, ολόψυχα, και ο Ευρωπαίος καταναλωτής σίγουρα καλύτερα θα ενημερώνεται με αυτή την ε, νομοθεσία. Ε, για μερικά προϊόντα. Κοιτάξτε αυτή την πίτσα που σας δείχνω με τυρί ε, από μπροστά η συσκευασία φαίνεται πολύ ε, ελκυστική. Από πίσω γράφει όμως ότι αυτό το τυρί ένταμ που λέει δεν είναι τυρί, είναι ε, νερό, ε, κάποια ίχνη τυριού, κρέμα και ε, φυτικά λίπη. Καλή σας όρεξη. Θα πρέπει παντού να γράφει λοιπόν τα προϊόντα υποκατάσταση. Βλέπω κύριε πίτροπε ότι νεύεται. στην πράξη τι κάνατε. Εγώ φοβάμαι στην πράξη θα γράφει σε αυτή την πίτσα ότι έχει φυτικά έλαια. Εντάξει, δεν τρομάζει ο καταναλωτής, σου λέει α, ωραίο είναι σαν, σαν ε, ελαιόλαδο και δεν καταλαβαίνει ότι είναι τεχνητό τυρί. Δεν μπορούμε το, το τυρί να γράφουμε τυρί και να, να γράφουμε ότι δεν είναι τυρί, μοιάζει με τυρί αλλά έχει αντικατασταθεί από φυτικά λίπη που έχουν όψη τυριού. Ε, χρειάζονται αυστηρή έλεγχη στα κράτη-μέλη τα ξέρετε κύριε Επίτροπε και σας προειδοποιώ, τα επόμενα χρόνια θα ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς εφαρμόζεται η παρούσα νομοθεσία στα κράτη-μέλη. Γιατί όπου γράφει τυρί θα πρέπει να έχει και μέσα τυρί. Αλλιώς θα πρέπει να το ξέρει ο καταναλωτή. Ελπίζω να πετύχει η εφαρμογή αυτή τη νομοθεσία. Αν δεν πετύχει, κύριε Επίτροπε, σίγουρα θα ζητήσουμε αυστηρότερη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Λάγκε. Για 1,5 λεπτό το λόγο έχει η κυρία Westlund. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ανήκω σε αυτούς ε, που είναι κατενθουσιασμένοι με το γεγονός ε, ότι έχουμε πια υποχρεωτική την επισήμανση για όλα τα είδη κρέατος για να γνωρίζουμε την προέλευση του κρέατος. Αυτό είναι σημαντικό και για τους καταναλωτές αλλά και για τους ε, γεωργούς και τους κτηνοτρόφους, γιατί στην ε, πατρίδα μου οι προδιαγραφές είναι πολύ υψηλότερες και αυστηρότερες. Ε, θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλιστούν συνθήκε ίσου ανταγωνισμού γιατί να μην έρθουν σε δυσμενή μεταχείριση δική μα γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Είναι καλύτερη για όλου αυτή η ρύθμιση, για το περιβάλλον, του καταναλωτέ και του γεωργούς. Επίσης, έχουμε διεύρυνση της υποχρέωσης αναφοράς χώρα προέλευση για πολλά προϊόντα. Δυστυχώς πολλές φορές οι καταναλωτές σήμερα παραπλανούνται από τις πληροφορίες που αναφέρονται στις ετικέτες. Χρειάζονται καλύτερη ενημέρωση και ευανάγνωστες πληροφορίες πάνω στις ετικέτες και ελπίζω αυτό να το καταφέρουμε στο εγγύς μέλλον. Βέβαια έχω και κάποια δυσφορία γιατί δεν δόθηκε αρκετή έμφαση στην ε, αναφορά των τρανς λιπαρών γιατί νομίζω ότι είναι καιρό να αποσυρθούν αυτά τα τρέσλι παρά από τι αγορέ. Επίση, για τα νανοηλικά θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η αναφορά στην επισήμανση. Και χαίρομαι για το ότι δεν πρέπει να δίνουμε πια το περιεχόμενο παρά ανά 100 γραμμάρια ή μιλιλίτρια. Έτσι θα μπορεί να κάνει πιο ενημερωμένα την επιλογή του ο καταναλωτής. Σας ευχαριστούμε κυρία Westland. Ο κύριος Τρεμός έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η τροπολογία 137 που καταθέσαμε με 40 άλλους συναδέλφους για τις γλώσσες στην επισήμαση ε, μιλάει για το σεβασμό της πολυγλωσσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το δικαίωμα των πολιτών να ενημερώνονται στη μητρική τους γλώσσα, ακόμη και αν η γλώσσα αυτή δεν είναι ακόμη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα η πολυμορφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ότι εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες έχουν μητρική τους γλώσσα, μία γλώσσα που δεν αναγνωρίζεται ως επίσημη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην περίπτωση Καταλανίας είναι πραγματικότητα ότι χιλιάδε χιλιάδες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την καταλανική γλώσσα για να, στις ετικέτες των προϊόντων τους εδώ και πολλά χρόνια και αυτό το έχουν επιδοκιμάσει εκατομμύρια καταναλωτές. Βέβαια, μερικές χώρες μπορεί να χρησιμοποιήσουν το άρθρο 52 για να ευνοήσουν οποιαδήποτε άλλη γλώσσα που δεν είναι ακόμη επίσημη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη το αίτημά μου και να δράσει αντίστοιχα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Όουσκι για ένα λεπτό. Thank you. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι μεταξύ εκείνων των Ευρωβουλευτών που έμειναν ικανοποιημένοι από το συμβιβασμό που επετεύθη. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία ε, Ζώμα, για το αποτέλεσμα αυτό της εξαιρετικής εργασίας. Μιλήσαμε για τη χώρα προέλευσης, για την ετικετοθεσία ιδιαίτερα στα προϊόντα κρέατος. Είναι λίγο ηρωνικό εξατμίζεται ο ενθουσιασμός ε, που θα μπορούσε κανείς να έχει για το κρέας να διαβάζει όλα αυτά. Θα πρέπει όμως ε, ο κανονισμός που εγκρίνουμε να είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών, αλλά δεν θα πρέπει να τους ε, καθοδηγούμε τους καταναλωτές να αποφασίζουν μόνοι τους και θα πρέπει να δούμε, μιλήσαμε για το ε, μέγεθος των χαρακτήρων πάνω στην ετικέτα, αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και το μέγεθο της συσκευασία κάθε φορά. Και να μην ε, επιβαρύνουμε περισσότερο ε, για τους καταναλωτές και όλο τον κλάδο. Εγώ θα ψηφίσω, εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστώ, ο πρόεδρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζει ότι ε, τα ξέρει όλα για τα πάντα, όλες τι ιστορίε και τώρα τα τρόφιμα. Αλλά ξέρετε, Βασιλιά είναι ο καταναλωτή και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο, ο ή οι καταναλώτρια επιλέγουν τι θέλουν να τρώνε. Βεβαίω, κάποιο είδο ε, ε, είναι κοινή λογική για τη διατροφική αξία ή τις αλλεργίες. Αλλά τα περισσότερα αυτά που λέει η τι αλλεργιε αλλα τα είναι υπερβολικά. Ε, και υπερβολικό ντάντεμα του καταναλωτή. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό ε, που ε, ζούμε μια οικονομική ύφεση. Και κάθε φορά που μιλάω τα ίδια λέω. Ξέρουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να ψηφίζει νόμους. Ε, το δικό μας κοινοβούλιο επί σειρά ετών ήταν γνωστό σήμερα η μητέρα όλων των κοινοβουλίων. Και αυτό είναι άλλο θέμα και άλλη μια απόφαση που θα πρέπει να λαμβάνεται σε επίπεδο κράτους μέλους. Ευχαριστώ. Κύριε Νούτα, το λόγο έχει για 1,5 λεπτό η κυρία Τάισεν. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, με τον κανονισμό αυτό, ο, κανονισμό, ο καταναλωτής επιτέλους έχει τις διατροφικές προφορίες που χρειάζεται για ε, να ε, ζει με τρόπο υγιεινό. Είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Ε, το γεγονό ότι ισχύει αυτό για όλα τα τρόφιμα πλέον και όχι μόνο εκείνα που φέρουν ισχυρισμού υγεία. Με ε, στάνταρ ποσότητες με αριθμητικά στοιχεία ε, η εναλλακτική λύση του φωτεινού σηματοδότη μπορεί να ήταν ελκυστική αλλά δεν ήταν ε, ικανοποιητική. γιατί επιβαρύνει πάρα πολύ ε, την παραγωγή και είναι σπάρος των ποιοτικών προϊόντων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και για τη νομοθεσία για τη γλώσσα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει δικαίωμα ενημέρωσης, αλλά τι να την κάνει την ενημέρωση όταν δεν την έχει σε γλώσσα που να καταλαβαίνει. Επίσης, υποστηρίζω ε, και τη διαφορά στο στόχο. Από τη μια ε, έχουμε την υποχρέωση για τη χώρα προέλευσης και από την άλλη την ε, υποχρέωση για ηχνή λασιμότητα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τα συστατικά να αναφέρονται από πού προέρχονται αργότερα. Αν αυτό είναι τόσο προβληματικό σήμερα, ας το αφήσουμε στην άκρη. Ευχαριστώ για ένα λεπτό ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάθε φορά που υπάρχει ένα συμβιβασμό χαιρόμαστε και προχωρούμε, αλλά δεν πιστεύω ότι ο συμβιβασμό αυτός είναι να τρελαθούμε από τη χαρά μας και να πέσουμε κάτω ξερή. Εντάξει, προχωρήσαμε σε ό,τι αφορά την επισήμανση των τροφίμων και ιδιαίτερα ε, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, την ποιότητα του μηνύματος, αλλά στα τρανς λιπαρά δεν προχωρήσαμε αρκετά, δεν είναι υποχρεωτική η σήμανσή τους και επίσης ε, θέλω να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην εξατλήσει τις προθεσμίες. Έχουμε τώρα προβλήματα ε, ε, υπέρβαρου, υπερβολικής κατανάλωσης τροφίμων την Ισπανία, στη Δανία, στην Αυστραλία έχουν ληφθεί μέτρα. Θα πρέπει να προχωρήσουμε και στην Ευρώπη. Καλή είναι η συμβασμή, αλλά θα πρέπει με σαφήνεια και με ε, προσοχή να τα ε, εφαρμόζουμε. Εντάξει, προχωρήσαμε, αλλά ας μην ξετρελόμαστε από τον ενθουσιασμό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Περεγιό. Για 1,5 λεπτό το λόγο έχει η κυρία Οκονή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχήν να επενέσω την εισηγήτρια για το έργο της. Είναι απαραίτητο κυρίε και κύριοι ο Ευρωπαίος καταναλωτής να έχει στη διάθεσή του στη συσκευασία ετικέτες που ε, δίνουν τι απαραίτητε πληροφορίες για το προϊόν ώστε να κάνει ενημερωμένο την ε, επιλογή του. Χαίρομαι για την συμβαστική λύση που βρήκαμε και δεν συμφωνώ με την ανάλυση του κ. Νάτχαλτ. Νομίζω ότι έχουμε λόγους να είμαστε ικανοποιημένοι γιατί οι πληροφορίες θα είναι πιο ευανάγνωστες, οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα θα είναι προσιτές στο κοινό, το ενδιαφερόμενο κοινό και οι απομιμήσεις θα αναφέρονται ως ε, ε, απομιμήσεις υποκατάστατα γιατί είναι απαράδεκτο να παραπλανούμε τον καταναλωτή πουλώντα ε, πουλώντας ένα τυρί που θα έχει γίνει από φυτικά αντί να έχει παρασκευαστεί από γάλα. Επίσης χαίρομαι που για τα κομμάτια κρέατος χοιρινού αγοπρόβιου ή πουλερικών αναφέρεται η προέλευσή τους στις συσκευασίες. Έτσι θα ενημερώνονται καλύτερα οι καταναλωτές και θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την περίπτωση μολύνσεων. Τώρα, για τι επιχειρήσει. Θα πρέπει σταδιακά να προσαρμοστούν στη, στο νέο κανονισμό. Αυτό προποθέτει κάποιε επενδύσει, αλλά και χρόνο για την προσαρμογή και τη συμμόρφωση με τι νέε διατάξει. Θα ήθελα λοιπόν να αφήσουμε το χρόνο σε αυτέ τι επιχειρήσει για να εφαρμόσουν αυτέ τι διατάξει χωρί να τροποποιούμε κάθε τρει και λίγο τον κανονισμό και επιβαρύνοντάς του όλο και περισσότερο. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό το λόγο έχει η κυρία Βερνιό. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πάνε τρία χρόνια που ασχολούμαστε με το θέμα αυτό και δεδομένου του δοκιμεύματο και τη τεράστια πίεση που μα ασκεί η αγροπιστική βιομηχανία, δεν μπορώ παρά να αισθάνομαι ικανοποιημένη από το αποτέλεσμά μα. Χαίρομαι ιδιαίτερω για την συμπερίληψη της, πλήρους, της υποχρεωτικής ετικέτας με την ε, θρεπτική και διατροφική αξία, ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να επιλέγει υγιεινά προϊόντα. Αναφέρονται πλέον σαφώς τα ελεργειογόνα, ακόμη και για τα μη προσκευασμένα τρόφιμα, και εξασφαλίζεται η αναγνωσιμότητα από το ελάχιστο μέγεθος της γραμματοσυράς. Επίσης, η υποχρεωτική μνήμα της προέλευσης, χώρας προέλευσης για όλα τα τεμάχια κρέατος είναι σημαντική και πολύ μεγάλη πρόοδος. Το ίδιο για τα, ε, για τα ψάρια και τα γάλα, τα, μετα, τα μεταποιημένα. Κρίμα. Ε, βέβαια χαίρομαι που το Ινόπνευμα δεν περιελήφθη γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστή ομοθετική διάταξη. Βέβαια θα μπορούσαμε να έχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα με ευανάγνωστη και εναρμονισμένη επισήμαση. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι κάναμε ένα σημαντικό βήμα για την καλύτερη ενημέρωση των Ευρωπαίων καταναλωτών. Ευχαριστώ κύριε Βερνιό. Για ένα λεπτό κύριο Σταμπάιτζη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι ε, κάτι θετικό ο συμβιβασμός αυτός, ε, εντάξει, αλλά μας απογοητεύει λίγο. Είναι προόδος να αναφέρεται σε όλα τα νοπά προϊόντα η χώρα προέλευσης. Καλό είναι αυτό. Αλλά λυπάμαι που δεν υιοθετήθηκε αυτό το σύστημα του φωτεινού σηματοδότη, το φανάρι. Ε, επίσης ε, η μερίσια ποσότητα και θερμίδες. Αυτό θα βοηθούσε πολύ περισσότερο τους καταναλωτές να τρέφονται με σωστό και υγιεινό τρόπο. Επίσης θα ενημέρωνε καλύτερα τους καταναλωτές σε μια ετικέτα στο πρόστιο μέρος της συσκευασία. Είναι ε, κάτι που δεν καταλαβαίνουμε. Ε, γιατί η δεξιά αντιτάχθηκε σε αυτό το μέτρο και δεν προχώρησε. Επίσης ήταν πολύ σημαντικό ε, για μένα να γράφουν και τα υνοπνευματόδηποτα ε, την ενέργεια που περιέχουν. Ευχαριστώ. Το λόγο για ένα λεπτό έχει ο κύριος ε, Ταραμπελά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ. Ε, σε αυτό το θέμα, πολύ περισσότερο από άλλο, η αρχή του «Καλύτερος είναι του καλού και ε, οι υπερβολικές ε, πληροφορίες, σκοτώνουν τις πληροφορίες, ε, ισχύει. Θα έπρεπε να έχουμε καλύτερες πληροφορίες. Χαιρόμαστε για την υποχρέωση μιας χώρας προέλευσης για όλα τα είδη και χαίρομαι για τη μάχη που δόθηκε και την κυρία Ρενάτα που το δέχτηκε. Βέβαια, η υποχρέωση μια χώρα προέλευση που μέχρι στιγμή ίσχυε μόνο για το βόλιο κρέα, το μέλι, το ελαιόλαδο, τα νοπόπορ και πευτικά, έχει τελικά επεκταθεί στο χείριο εγωπρόβιο και κρέα πουλερικών σε νοπή κατάσταση. σω θα έπρεπε να επεκτείνουμε αυτή την υποχρέωση και σε άλλα τρόφιμα. Βέβαια, η συμβαστική αυτή λύση δεν ικανοποιεί πλήρω όλου του καταναλωτέ, αλλά ήταν δύσκολη η επίτευξη ακόμη και αυτή. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει συμπληρωματικέ διατάξει το συντομότερο δυνατό, χωρί όμω να έχουμε επαχθεί μελέτε. Και γιατί να προσδιορίσουμε τη μερίδα, δεν σα ζητάμε να προσδιορίσετε τη μερίδα, να αναφέρεται η περιεκτικότητα 100 γραμμάρια η μιλιλίτρ και όταν υπάρχουν ε, ξεχωριστά, ε, ξεχωριστές μονάδες αναφέρεται. Η μερίδα δεν έχει πια νόημα να αναφέρεται γιατί δεν υπάρχει εναρμονισμένη μερίδα. Ευχαριστώ κύριε Ταραμπέλα. Τώρα περνάμε στη διαδικασία του Catch the Eye. 13 ε, βουλευτές ζήτησαν το λόγο. Και έχουμε ήδη μείνει λίγο πίσω, αρκετά μάλλον πίσω. Γι' αυτό δεν θα δω το λόγο και στους 13. Θα δώσω το λόγο μόνο σε 6 ευρωβουλευτές προσπαθώντας να κάνω μια ισορροπημένη κατανομή μεταξύ των πολιτικών ομάδων και φυσικά τηρώντας ε, τη σειρά με την οποία εγγραφήκατε. Το λόγο έχει για ένα λεπτό κύριο Σκέλη. Ε, Οι περισσότεροι βουλευτές ε, χαιρετίζουν αυτές τις προτάσεις και αυτό εντυπωσιάζει γιατί βοηθάει τους καταναλωτές ε, και ε, πρέπει να έχουμε κατά νου το ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, δεν θα πρέπει να εξαφανιστούν και να επικρατήσουν οι πολυεθνικές. Πρέπει να πω με μεγάλη μου χαρά, μπόρεσα σήμερα το πρωί να έχω πρωινό με μια ομάδα γυναικών που μου ανέφεραν τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήγαγαν οι περισσότεροι αισθάνονται ότι είναι απαραίτητο να φέρεται η ένδειξη της προέλευσης και πάνω από 50% όσων απάντησαν δεν γνώριζαν ότι η ετικέτα με την ένδειξη προέλευσης σημαίνει κατ' ουσίαν τη χώρα όπου έγινε η τελευταία σημαντική αλλαγή. Υπάρχει όμως μια μεγάλη διαφορά από το αν κάτι έχει παραχθεί στη χώρα ή έχει μεταποιηθεί στη χώρα. Άρα δηλαδή πρέπει αυτό να διευκρινίζεται. Ευχαριστώ κύριε Κέλλη. Το λόγο τώρα έχει για ένα λεπτό ο κύριος Τσέμκε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτρια και χαίρομαι για πρώτη φορά, που για πρώτη φορά στη συζητήση μας στην αίθουσα αυτή συμμετέχει και ο Υπουργός Σαβίτσκι και θα ήθελα να τον καλωσορίσω. Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και πολύ συχνά Μιλάμε εδώ για τις υποχρεώσεις των παραγωγών. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο εξής. Αυτές οι συστάσεις είναι πολύ σημαντικές για τους καταναλωτές και οι καταναλωτές χάρη στις πληροφορίες αυτές θα ενημερωθούν καλύτερα και θα γνωρίζουν καλύτερα τα δικαιώματά τους. Βέβαια αυτό είναι ο σκοπό, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα ενημερωθούν ε, σίγουρα οι καταναλωτέ. Είναι σημαντική να γίνει μια διαπαιδαγώγηση των καταναλωτών, γιατί δεν αρκεί να έχουμε περισσότερα στοιχεία και περισσότερε πληροφορίε στι ετικέτε. Το σημαντικό είναι να ενημερώνονται όχι μόνο οι δίκοι, αλλά και οι απλοί καταναλωτέ να μπορούν να διαβάζουν τι πληροφορίε και να κατανοούν τι πληροφορίε που περιλαμβάνονται στι ετικέτε. Σα ευχαριστούμε κύριε Ζέμκε. Για ένα λεπτό έχει το λόγο ο κύριο Όμπερμαϊερ. Κύριε Πρόεδρε, έχουν περάσει τρία χρόνια και πολλά σκάνδαλα για να βρούμε ένα συμβιβασμό. Έχουμε γάλα, που, ε, κρέας που δεν γίνεται από γάλα, ε, το ε, ζαμπόν, το λουκάνικο που είναι από διάφορα υπολείμματα. Αυτό όμως δεν είναι δυνατόν να προσφέρεται στον καταναλωτή. Βεβαίως η προέλευση, ούτε και αυτή είναι ικανοποιητική, η ένδειξη προέλευσης κρέατος και θα πρέπει να υπάρχει ένδειξη και για μεταποιημένα προϊόντα αν αυτά έρχονται από την Βραζιλία ή από την Τελάντη και για το ε, προσούτο πρέπει να πούμε ότι αυτό συνήθως ε, δεν έρχεται από τη γνωστή περιοχή αλλά πολύ βορειότερα. Η έκθεση αυτή λοιπόν έπρεπε εδώ και πολύ καιρό να γίνει, έγινε προς σωστή κατεύθυνση, πρέπει όμως να παραμείνουμε στάσιμοι και να περιμένουμε το επόμενο σκάνδαλο για να δραστηριοποιηθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τώρα για ένα λεπτό η κυρία Ροτ Πέρεντ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θα επιθυμούσα οι συνάδελφοι να ήταν πιο θαραλέοι και να είχαν τολμήσει μια δεύτερη ανάγνωση και μια συνδιαλλαγή ανεξάρτητα από την Προεδρία. Δεν έχουμε ετικέτα στην πρόσθεια ε, όψη, ούτε καν αναφέρονται οι θερμίδες, ούτε οι θερμίδες στο ενόπνευμα, για να μην πω για άλλες ε, ουσίες, ε, ούτε πόσο είναι η θερμίδα, ό,τι και να είναι. ένα κουτάλι, ένα φλιτζάνι, η μερίδα, συγγνώμη. Η, χώρα προέλευσης, κάτι που θέλουν να γνωρίζουν επιγόντως οι καταναλωτές, δεν ρυθμίζεται σωστά και ε, στο άρθρο 25 ε, ε, θέτουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το ψάξει τα τρανς λιπαρά, τα συστατικά. Αυτά είναι πρώτης και δεύτερης τάξεως κηδεία, δεν δείχνουν θάρρος και σθένος. Ας πηγαίναμε στη δεύτερη ανάγνωση και στη συνδιαλλαγή να είχαμε ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα. Έτσι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές δεν μπορούν παρά να μείνουν απογοητευμένοι. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει για ένα λεπτό ο κύριος Ντόρφμαν. Danke, Herr Präsident. Ich glaube, wir haben Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι επιτύχαμε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτρια. Νομίζω ιδιαίτερα το άρθρο 9, όπου πρόκειται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι ένα σημαντικό άρθρο σε πάρα πολλές περιοχές της Ένωσης τα τελευταία χρόνια. Έχουμε άμεση εμπορία, προωθήσαμε την άμεση εμπορία από αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει τώρα να μεριμνήσουμε να μην επηρεαστούν τέτοιου είδους εμπορικές δραστηριότητες. Βεβαίως όσον αφορά τα αλκοολούχα ποτά θα ήθελα να είμαστε λίγο πιο θαραλέοι. Νομίζω είναι κατανοητό ότι για τα αλκοπόψ ε, θα πρέπει να προβλέπεται η επισήμανση. Για το κρασί ε, θα μπορούσαμε να επιτύχουμε μια μακροχρόνια εξαίρεση έχοντας κυρίως κατά νου ότι εδώ και δεκαετίες για το κρασί ισχύουν διατάξεις ε, οι οποίες είναι πολύ πιο αυστηρές από ό,τι για άλλα προϊόντα Παραδείγματο χάρη για το κρασί πρέπει να αναφέρεται περιεκτικότητα πνεύματο, ε, προέλευση, ε, μέγεθο, ποσότητα. Νομίζω λοιπόν ότι ε, στο μέλλον δεν πρέπει να αλλάξουμε τίποτα, τίποτα όσον αφορά τι ενδείξει για το κρασί. Η κυρία Μάνερ, παρακαλώ. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πολύ ε, καλή ικανοποιητική συμβασική πρόταση που είναι οπωσδήποτε ένα βήμα προς τα εμπρός. Όταν μιλάμε για την επισήμανση είναι σαφές ότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου κυρίως ε, τον καταναλωτή και τα δικαιώματα του καταναλωτή. Ο καταναλωτής ε, πρέπει να γνωρίζει τι περιέχει το προϊόν το οποίο αγοράζει και βεβαίως πρέπει να υφίσταται η δυνατότητα να προτιμώνται τα τοπικά προϊόντα. Ε, κατόπιν τούτου η σήμανση προέλευσης είναι πολύ σημαντική και πρέπει αυτή να επεκταθεί ε, και σε άλλα είδη κρέατος. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως ε, υπολείπονται ακόμα πολλά αλλά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα παραδείγματο χάρη και τα μεταποιημένα προϊόντα και αυτά ε, πρέπει να συμπεριληφθούν περισσότερο έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση. Κατά τα άλλα συμφωνώ πολύ με αυτό που είπε ο κύριος Τρίμοζα. Ευχαριστώ. Τελευταία τοποθέτησε ο κύριος Μικολάση για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα για το πώς μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βοηθήσει επικοδομητικά έτσι ώστε ε, να βοηθήσουμε τους πολίτες σε ένα θέμα που τους ενδιαφέρει και που καταλαβαίνουν. Χαίρομαι για αυτό που αποφασίσαμε για την ενημέρωση, για το μέγεθος της γραμματοσυράς. Ως γιατρός επίσης χαίρομαι που θα αναγράφονται διάφορες ουσίες, αλλεργιογόνα και άλλες που ε, προκαλούν προβλήματα ανοχής ή δυσανεξίας. Μπορούμε να δούμε, ας πούμε, ε, μια ετικέτα με ωραίες φράουλες και μέσα το προϊόν να έχει κάποια τεχνητά υποκατάστατα και καμία σχέση με φράουλες. Χαίρομαι κύριε Επίτροπε που αναφέρατε και άλλα θέματα για το μέλλον, ε, για τις θερμίδες, για τα εινοπνευματόδια, ότι θα τα μελετήσετε και θα κάνετε προτάσεις στο μέλλον για να βελτιωθεί τόσο καλή έκθεση κυρίας Ρενάτε Σόμερ. Την ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Ο Πρόεδρος. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Επίτροπος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους βουλευτές. Είναι κρίσιμο να πούμε και να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλει και μπορεί να παράγει νομοθεσία που πραγματικά ενισχύει ε, τους πολίτες στην καθημερινή τους ζωή και ε, για να έχουν δύναμη στα χέρια τους οι πολίτες θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι. Συμφωνώ με τον κύριο Γκερμπράντη που είπε η βελτίωση της τεχνολογίας στο μέλλον θα μας επιτρέψει να είμαστε ε, πιο χρήσιμοι στους καταναλωτές και να τους ενημερώνουμε γέρος για το τι ε, καλούνται να καταναλώσουν. Σημείωσα την επιμονή ορισμένων βουλευτών στο θέμα της εφαρμογής και της επιβολής νομοθεσίας. Αναφέρατε επίσης και το θέμα της φαγής των ζώων χωρίς αναισθησία ή το θέμα των διαφόρων απομιμήσεων. Πάντα τονίζατε την υπόθεση της εφαρμογής. Αυτό είναι πραγματικά το κλειδί. Πιστεύω ακράδαντα ότι ακόμα και πριν φέρουμε νέους κανόνες και νέα νομοθεσία, νέους κανονισμούς, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι αυτά που σήμερα ισχύουν εφαρμόζονται σωστά. Και πιστεύω ότι οι προσπάθειες που κάνουμε και οι πόροι που αφιερώνουμε θα πρέπει όλο και περισσότερο να είναι στοχευμένοι προς την κατεύθυνση αυτή της ε, εξασφάλισης της υλοποίησης. Επίση θα πρέπει να είμαστε πολύ δημιουργικοί στην απομίμηση. Συμφωνώ με την κυρία Ντελάγκε, διότι ενώ δίνουμε τη σωστή πληροφόρηση στους καταναλωτές ως προς την παρουσία ή την απουσία ορισμένων ουσιών σε ένα προϊόν, δεν θα πρέπει να δίδεται η ευκαιρία, πώς να το πω, δημιουργικού μάρκετινγκ να χρησιμοποιούν τον κανονισμό μας εις βάρος μας τονίζοντας το προϊόν ότι και λέγοντας, πούμε, με μικρότερη γραμματοσυρά ότι είναι άλλο. Θα πρέπει και εμείς να είμαστε πάρα πολύ εφάνταστοι και δημιουργικοί όταν κάνουμε τον κανονισμό αυτό. Συμφωνώ με την κυρία Λεωτάρνη, είμαι και εγώ πολύ απογοητευμένος που δεν έχουμε ε, για την κλωνοποίηση κανονισμό, ούτε ενημέρωση για την κλωνοποίηση των ζώων. Χάσαμε την ευκαιρία, πιστεύω, να μπούμε στο, δρόμο ε, για την ενημέρωση αυτή στο μέλλον. Πιστεύω ότι οι προτάσεις που είχαμε σήμερα, ή μάλλον πριν από μερικές εβδομάδες, χωρίς να είναι η τελική στόχη, που έχουμε περισσότεροι στο μυαλό μας, εν πάση περιπτώσει μας δείχνουν την κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να κινηθούμε έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια θέση όπου θα δίδεται αυτή η πληροφόρηση στους καταναλωτές για να ξέρουν τι καταναλώνουν. Αυτό είναι το κλειδί, εν πάση περιπτώσει. Θυμάμαι, ε, κατά τη διάρκεια της ακρόασης μου στο Κοινοβούλιο, είχα δηλώσει με τρόπο κατηγορηματικό το θέμα είναι όχι να λέμε στον κόσμο τι να φάει, αλλά να, πούμε στον κόσμο τι τρώει και να αποφασίσει τι θέλει πραγματικά να κάνει. Στο θέμα των γλωσσών και πάλι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν αλλάξαμε τον ισχύοντα κανονισμό για τις γλώσσες. Και θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί, αν κατάλαβα καλά, η τροπολογία που προτείνεται θα επέτρεπε σε οποιαδήποτε χώρα, περιφέρεια, η επαρχία να επιβάλλει μία αποκλειστική γλώσσα ε, στη συσκευαστία. Και πάλι αυτό δεν εξυπηρετεί το στόχο της ενημέρωσης. Δεν βελτιώνει την πληροφόρηση των καταναλωτών. Η νέα νομοθεσία αποτελεί ορόσημο στα δικαιώματα του Ευρωπαίου καταναλωτή στην ενημέρωση με την νομοθετική διαδικασία που ολοκληρώνεται μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη φάση της εφαρμογής. Απομένει βέβαια ακόμα πολλή δουλειά να γίνει για να βεβαιωθούμε ότι θα εφαρμόζονται πλήρως ορισμένοι κανόνες. Προσβλέπω στην πλήρη διοργανική συνεργασία για να εξασφαλίσουμε τη σωστή εφαρμογή και υλοποίηση αυτή τη νομοθεσία. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω την εισηγήτρια δόκτωρα Σόμερ και του και για τι προσπάθειε του που ήταν μεγάλε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Το λόγο έχει τώρα εκ μέρους του Συμβουλίου ο κύριος Σαβίτσκι. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ, η συζήτηση κράτησε πάνω από τρία χρόνια και ακόμη έχουν απομείνει πολλές αφιβολίες και ε, μια διακύμανση των απόψεων από αμέριστη υποστήριξη, επιφυλάξεις μέχρι μεγάλη απογοήτευση όπως εξέφρασε ο Ευρωβουλευτής κύριος Σταμπάιτζη. Κυρίε και κύριοι, το τι τρώμε ουσιαστικά προσδιορίζει και τον τρόπο ζωής μας και φυσικά ως καταναλωτές έχουμε δικαίωμα για σωστή ενημέρωση για τα τρόφιμα που καταναλώνουμε γιατί δεν θα πρέπει ε, να κάνουμε διατροφικά λάθη. Δεν θα πρέπει να κάνουν διατροφικά λάθη ε, οι συνάδελφοι του κυρίου Μικολάησικ. Πριν από λίγο ακούσαμε την ομιλία του Επιτρόπου Ντάλι. Ο Επίτροπος μας είπε ότι οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να, να πληροφορηθούν από μας τι πρέπει να φάν, αλλά έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τι είναι αυτό που τρώνε. Και από την ε, ετικέτα μόνο δεν μπορούμε ε, να διαπαιδαγωγήσουμε τους καταναλωτές και να δημιουργήσουμε καλές διατροφικές συνήθειες. Δεν αρκεί μόνο μία ετικέτα, δεν αρκεί μία μόνο μία σωστή επισήμανση. Χρειάζεται μία τεράστια προσπάθεια ενημερωτική, μία διαπαιδαγώγηση του καταναλωτή. Δυστυχώς μόνο η επισήμανση του προϊόντος δεν αρκεί για αυτή τη διαπαιδαγώγηση και τη σωστή ενημέρωση. Συμφωνώ με τον Επίτροπο Ντάλι ότι αυτό που έχουμε σήμερα με τη μορφή συμβαστικής πρότασης είναι μια εξισορρόπηση μεταξύ των προσδοκιών και των συμφερόντων του καταναλωτή και των δυνατοτήτων των παραγωγών, των γεωργών και των μεταποιητών της μεταποιητικής βιομηχανίας. Θα ήθελα να επισημάνω το ζήτημα της σφαγής, της ευημερίας των ζώων, το θέμα της κλωνοποίησης των ζώων, το σχόλιο που έκανε η κυρία Λιωτάρ και για τα σημεία αυτά θα πρέπει στο μέλλον να υπάρξουν διευκρινήσεις και συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις. Αναφέρατε συγκεκριμένα στην ε, ανάγκη και υποστηρίξατε την υποχρεωτική μνήμα της χώρας προέλευσης. Θυμάμαι τις συζητήσεις που έγιναν στην προηγούμενη διεύρυνση το 2004 όταν οι νέες χώρες μέλη με σαφή τρόπο έλαβαν την πληροφορία ότι η μνήμα της χώρας προέλευσης ε, ε, ισοδυναμεί ουσιαστικά με εμπορικό προστατευτισμό. Αυτό είχαμε ακούσει. Αλλά χαίρομαι που στη διευρυμένη σήμερα Ευρώπη αναγνωρίζουμε ότι οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα στη γνώση, έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν την προέλευση των προϊόντων που αγοράζουν. Και πραγματικά αξίζει να ε, έχουμε σωστή επισήμανση και των εξοκοινωτικών προϊόντων. Γιατί τα προϊόντα που παράγονται και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τηρούν τι ίδιε υψηλέ προδιαγραφέ με τα προϊόντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει και το θέμα αυτό να το συζητήσουμε. Επίση, πολύ σημαντικό είναι το ζήτημα τη απομίμηση των προϊόντων. Γιατί δυστυχώ αυτή η διαδικασία είναι αρκετά ε, εκτεταμένη, διαδεδομένη και δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε. Είναι πολύ σημαντικό αν ένα προϊόν είναι ζωικής προέλευση ή όχι. Θα πρέπει να ξέρουμε ένα προϊόν, ένα συστατικό είναι υποκατάστατο. Θα πρέπει όλα αυτά να αναφέρονται στην ετικέτα ώστε να γνωρίζουν ε, οι καταναλωτές με ακρίβεια τι ακριβώς αγοράζουν, τι καταναλώνουν. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση και να σας διαβεβαιώσω ότι όλες σας οι ανησυχίες και οι φόβοι θα διαβιβαστούν από μένα στο αρμόδιο Υπουργικό Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σαβίτσκι. Για να ολοκληρωθεί η συζήτηση, το λόγο έχει τώρα η συγγήτρια κυρία Σόβα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κοιτάξτε αγαπητοί φίλοι, όλοι θα θέλαμε κάτι παραπάνω. Όλοι είχαν πολύ ωραίες ιδέες και εγώ ε, θα ήθελα η ένδειξη θερμίδων να είναι υποχρεωτική στο, στην συσκευασία, ανακατογραμμάρια ή οτιδήποτε άλλο. Και άλλοι είχαν και άλλες επιθυμίες, αλλά βάση πάση περιπτώσει όταν επιθυμούμε το συμβασμό θα πρέπει να υποχωρήσουμε και Ίσως αυτό ε, να σας αρέσει, ίσως και όχι, αλλά μόνο έτσι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια λύση. Εγώ λοιπόν δεν θεωρώ ότι είναι σωστό σε ένα τόσο δύσκολο θέμα να ε, ζητάμε τη συνδιαλλαγή. Γιατί όποιος τη ζητά τη συνδιαλλαγή και αυτό το ζητάει η τροπολογία που θα ψηφιστεί αύριο, όποιος λοιπόν επιθυμεί την ε, διαπραγμάτευση θέλει να καταστρέψει κατ' ουσίαν τη συμβαστική πρόταση που έχουμε επιτύχει γιατί είναι σαφές ότι στη διαπραγμάτευση ε, θα αποφασίσει αυτό το θέμα ακριβώς όπως απέτυχε πρόσφατα και ο κανονισμός για τα νέα τρόφιμα. Κατόπιν τούτου όλοι οι συγητές των πολιτικών ομάδων συνέβαλαν στο να επιτύχουμε αυτό που πετύχαμε και συμβάλλεται και εσείς αγαπητοί συνάδελφος Λιωτάρ εκ μέρους της Γκουε και ο κύριος Ρώση για τη δική του την πολιτική ομάδα. Γι' αυτό λοιπόν δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν τώρα να αποσύρεστε από τη συμβαστική πρόταση και να λέτε μα αυτό που προέκυψε είναι ένα τερατούργημα και εμείς δεν μπορούμε να το στηρίξουμε, δεν αρκεί. Ε, τότε αν είναι έτσι γιατί είχατε συμφωνήσει καταρχήν εσείς είχατε βοηθήσει να ε, συμπήξουμε αυτό το συμβασμό και γι' αυτό και ευγνώμονος. Ε, δηλαδή, κατ' ουσίαν τι λέτε, λέτε ε, πλύνε με αλλά μην με βρέξει. Αυτό όμω είναι λαϊκίστικη προσέγγιση. Δεν είναι σωστό. Θέλουμε να κάνουμε κάτι για τον καταναλωτή κάτι το σημαντικό για τον καταναλωτή. Δεν είναι τέλειο, προφανώς και θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Αντιαμφισβήτητα Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να επιλύσουμε στη μεταβατική περίοδο μέχρι τελικά να εφαρμοστεί αυτός ο κανονισμός. Όμως εγώ ε, νιώθω μισοσύνη για την Επιτροπή ότι θα βρει τη λύση και πράγματι θα διεξάγει έρευνε για θέματα εινοπνεύματος ότι θα δώσει τον ορισμό του αλκοπόψ. Ε, θα καταλήξουμε πιστεύω σε πολύ καλή λύση και γι' αυτό επιθυμώ αύριο να στηρίξετε αυτόν τον πολιτικό συμβασμό. Ευχαριστούμε κυρία Σόμερ. Ολοκληρώνουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Η ψηφοφορία του θα γίνει αύριο στις 12.30. Περάμε στο επόμενο σημείο της ημέρης διάταξης την έκθεση Ροτ Βέρεντ για την ομοθεσία